Bene, allora cominciamo i lavori della Commissione di oggi pomeriggio. Ξεκινάμε τις απομερινές μας εργασίες στο σημείο 21. Α, πριν πάμε στα σημεία, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το τι έγινε στην συνεδρίαση των συντονιστών που αποφάσισαν στις 6 Σεπτεμβρίου οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τα ονόματα των βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία της Ιρλανδίας ε, προτάσεις για τις μερίδες μελέτης για το 2013, τις απόψεις του όσον αφορά το σχέδιο των συνεδριάσεων για το 2013, για τις αντιπροσωπείες για το 2013, για τις δημόσια ακροάσεις του 2013 και για τις ιδέες που έχουν ενδεχομένε για ενδεχόμενε συναντήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ενεκρίθη εξάλλου το πρόγραμμα των δημοσίων ακροάσεων για το χάρτη πορείας μέχρι το 2050. Ακροάσει όσον αφορά τις αρμοδιότητες της ΙΤΡΕ, όσον αφορά την εξεργασία των στοιχείων. Μία ενημέρωση, ένα briefing όσον αφορά ε, την, ε, την καινοτομία Ευρώπη, Αμερική και επίσης τεχνολογική συνεργασία με την ε, Βραζιλία που αφορά εμένα. Αυτά συνοπτικά ήταν ε, αυτά που αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών χθες το βράδυ. Όσον αφορά όμως τα σημερινά, συστήματα, συγγνώμη, τα σημερινά θέματα της σημερινής διάταξης και το πρώτο σημείο τη συναδέλφου Πιλάρ Δεκαστήγιου, η οποία κανονικά θα έπρεπε να παρουσιάσει την έκθεση τη αντιπροσωπεία που μετέβη στη Βραζιλία. Ενημέρωση. Δεν μπορούσε να παρίσταται το απόγευμα και έστειλε σε όλου του βουλευτέ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Επιτροπή Ήτρε την ενημέρωση αυτή. Την έκθεση. Οπότε και το σημείο 21 ε, το έχουμε κάνει. Έχουμε τρία σημεία ακόμα στην ημερήσια διάταξη, το 22, το 23 και 24. Επ' αυτών θα να ακούσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις θα ακουστούν. Στο τέλος ε, θα ζητήσουμε. Δίνω το λόγο όμως αμέσως για το πρώτο σημείο. Διαδικασία αδειοδότησης για το πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα. Έχετε το λόγο, εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ στο Κοινοβούλιο σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Θέλουμε σήμερα να εστιάσουμε στο φάσμα για τις τεχνολογίες 4G. Αυτή η τεχνολογία και ιδίως η τεχνολογία DLT η οποία αναφέρεται πάντα σε σχέση με το πρόγραμμα με το σύστημα 4G, δηλαδή τετάρτης γενιάς, θεωρείται από το Κοινοβούλιο ως ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορούμε να έχουμε <clears throat> υπηρεσίες διαδικτυακές υψηλού επίπεδου σε κινητά τηλέφωνα, επομένω και στου πολίτε. Για να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο ο οποίο είναι αποτελεσματικό σε σχέση με τη χρησιμοποίηση του ραδιοφάσματο, κάτι το οποίο θα μα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα έλλειψη χωρητικότητα λόγω του υψηλού ρυθμού μετάδοση δεδομένων και για την καλύτερη χρησιμοποίηση του ραδιοφάσματο για άλλε ε, σημαντικές υπηρεσίες που έχουν ενδιαφέρον για του πολίτε. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο ενεκρίθη από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο αυτού του έτους έχει εστιάσει στη χρήση του ραδιοφάσματος για ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητού χαρακτήρα. Ένα βασικό στοιχείο στο οποίο έχει δώσει μεγάλη έμφαση το Κοινοβούλιο στο έργο του είναι να καλύψει να αποφασίσει για μια περιοχή 12.200 MHz εύρους φάσματος που θα ήταν ελεύθερη από άλλες χρήσεις και αυτό σχετίζεται με το, κατά κάποιο τρόπο, με το στόκ για το ραδιοφάσμα το οποίο έχει αναλάβει να κάνει η Κομισιόν για τον απολογισμό για το, της χρήσης του φάσματος. Αλλά ιδιαίτερα για την ασύρματη τις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις μέσα στο πρόγραμμα αυτό σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες εναρμονισμένες περιοχές ραδιοφάσματος, σε δύο μορφές πρώτα απ' όλα. Σε ό,τι αφορά το ραδιοφάσμα το οποίο έχει τύχη τεχνικής εναρμόνισης, δηλαδή έχει ήδη εντοπιστεί ως χρησιμοποιούμενο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ασύρματη ασύρματε ευρωζωνικέ υπηρεσίε, που είναι το αντικείμενο τη απόφαση τη Κομισιόν, τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση μέχρι το τέλο του 2012 να δώσουν τι ε, αδειοδοτήσει για τη χρήση αυτών των ε, περιοχών φάσματος. Δεν θέλω να γίνω ιδιαίτερα τεχνικός. Το Κοινοβούλιο παρόλα αυτά κατάλαβε όλα αυτά τα οποία ε, διακυβεύονται. Υπάρχουν τέσσερις ε, ζώνες, 900 MHz, 800 MHz, 2,6 GHz και 3,6 GHz είναι οι τέσσερις ζώνες και υπήρξαν το αντικείμενο τεχνικής εναρμόνισης εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμιά περαιτέρω δικαιολογία για να καθυστερήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης, ώστε οι πάροχοι ευρυζωνικών κινητών υπηρεσιών μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Έχουμε περίπου 870 MHz εύρους ζώνη για ασύρματες ε, ευρυζωνικές ε, επικοινωνίες αυτή τη στιγμή. Θα σας δώσω και περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την πρόοδο στα κράτη-μέλη για την αδειοδότηση Υπάρχει επίσης μια πρόσθετη <clears throat> υποχρέωση για τη ζώνη των 800 MHz, η οποία αναφέρεται ως η ζώνη του ψηφιακού μερίσματος, γιατί προηγουμένως χρησιμοποιείται για αναλογικές εκπομπές τηλεόρασης και από τότε που έχουν περάσει σε ψηφιακή εκπομπή τα τηλεοπτικά κανάλια, αυτό το τμήμα του φάσματος είναι ελεύθερο για άλλες χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι και πάλι είχαμε μια διαδικασία τεχνητή, τεχνικής εναρμόνισης για να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό την ε, ζώνη για ευρυζωνική ασύρματη επικοινωνία. Τελικά, λόγω τη πολιτική σημασία, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ήταν αυτό που, αυτά που έπρεπε να αποφασίσουν για αυτά και αυτό κάνετε με το πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα πρέπει να έχει περατωθεί η διαδικασία αδειοδότησης για την ζώνη των 800 MHz. Είναι υποχρεωμένα λοιπόν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στη διαδικασία αυτή αδειοδότηση, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η περιοχή του φάσματο για βριζονικέ ασύρματε υπηρεσίε. Επίση, θέλω να σα δώσω κάποιε πληροφορίε για αυτά που γνωρίζουμε σε σχέση με την πρόοδο στα κράτη-μέλη για αυτή τη ζώνη του φάσματο. Αφού όμω προηγουμένω δούμε το σύνολο όλων αυτών των ζωνών που έχουν απελευθερωθεί και έχοντα υπόψη του κύριου στόχου που έχει θεσπίσει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την απελευθέρωση των 1200 ε, MHz σε εύρος φάσ, ε, φάσματος για ευρυζωνικές ασύρματες υπηρεσίες, είναι σαφές ότι έχουμε δει καταστάσεις όπου τα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να αναλάβουν τις τεχνικές αποφάσεις εδώ και πολύ καιρό, εξακολουθούν να χρονοτριβούν και να καθυστερούν σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Και επιπλέον, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή τηλεόραση και τη μετάβαση από αναλογικές σε ψηφιακές εκπομπές που οδηγούν σε προβλήματα για ορισμένα κράτη-μέλη και η χρήση στρατιωτικών τεχνολογιών καθιστούν αυτή τη διαδικασία. Διαδικασίες λοιπόν που εκκρεμούν ακόμα σε ορισμένα κράτη-μέλη και επομένως σε σχέση για τις τέσσερι εναρμονισμένες ζώνες του φάσματος που ανέφερα προηγουμένως, ξέρουμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν περατώσει την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών στην εθνική νομοθεσία και όλα τα κρατημέλη, από ό,τι γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί, έχουν περατώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο, ιδίως για την ανακατανομή και την αναπροσαρμογή της ε, ζώνης των 800 MHz που ήταν στο παρελθόν η ζώνη, όπως τη λέγαμε, GSM, αλλά το Κοινοβούλιο είχε εμπλακεί πλήρω σε αυτή τη διαδικασία να εξασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιείται αυτή η ζώνη για πιο σύγχρονε καινοτόμε τεχνολογίε. Αλλά δυστυχώ παραμένουν ορισμένε καταστάσει όπου κράτη-μέλη δεν έχουν αδειοδοτήσει αυτέ τι ε, ζώνε. Στην ζώνη των 2,6 GHz μόνο τα μισά κράτη-μέλη έχουν περατώσει τη διαδικασία αδειοδότηση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 7 ακόμα κράτη-μέλη τα οποία είναι ενεργά εμπεπλεγμένα στην διαδικασία αδειοδότησης ή την έναρξη αυτής της διαδικασίας και τους πληστηριασμούς για ορισμένε ζώνες, αλλά ξέρουμε ότι αυτά τα κρατη δεν θα έχουν περατώσει τη διαδικασία στο τέλος του χρόνου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτή η ζώνη έχει συνδεθεί από τους παρόχους υπηρεσιών και από τους τεχνολογικούς υπευθύνους ως μια ζώνη η οποία δουλεύει πολύ καλά ε, χέρι-χέρι μαζί με τη ζώνη των 800 MHz, δηλαδή 2,6 και 800. Στο παρελθόν η ζώνη των 900 MHz για τα GMSM είχε συνδεθεί με τη ζώνη 1800 ε, MHz, τώρα τα 800 MHz πάνε μαζί με τα 2,6 GHz χέρι-χέρι. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι και οι δύο ζώνε θα απελευθερωθούν παράλληλα, ώστε να έχουμε κοινέ υπηρεσίε οι οποίε θα μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα 800 MHz τη ζώνη αυτή, αυτήν κάθε αυτήν, σε 7 κράτη-μέλη έχει τύχει πλήρου αδειοδότηση. Υπάρχουν επίσης και εξελίξεις για την αδειοδότηση σε άλλα 7 κράτη-μέλη, δυστυχώς όμως. Σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και εκεί καθυστερεί η διαδικασία. Τρία ακόμα σχεδιάζουν να μπουν σε διαδικασίες αδειοδότησης για του χρόνου, το 2013 δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε τουλάχιστον άλλα 7 κρατη όπου δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη ότι θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με κάποια σπουδή. Αλλά το πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα αναγνώρισε το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν ορισμένα κράτη-μέλη προβλήματα, ιδίως στα κράτη-μέλη όπου χρειάστηκε να, αποτραπεί, να αποτραπούν παρεμβολές με συστήματα αεροραδιοπλοήγησης παραγωγή χάρη χώρες όμω με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και εκεί υπήρξε καθυστέρηση τη προόδου για τη χρήση τη ζώνη του, των 800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικέ υπηρεσίε. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει διαπραγματεύσει και έχουν περατωθεί διμερεί συμφωνίε μεταξύ μερικών κρατών μελών τη Ρωσία και τη Ουκρανίας και από ό,τι βλέπουμε λοιπόν δεν υπάρχουν, ακόμα πραγμα... δεν υπάρχουν πια πραγματικά προσκόμματα για να μπορέσει να περατωθεί αυτή η διαδικασία διοδότηση στι χώρε αυτέ. Παραμένουν όμω ανησυχίε σε σχέση με παρεμβολές για τα, από τα τηλεοπτικά κανάλια. Ξέρουμε ακόμα ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεκκλήσεις για 7 χώρες. Ήδη δύο κρατημέλη έχουν ζητήσει μια παρέκκληση, έχουν αναφέρει ότι για ρόους που έχουν εξηγήσει δεν θα μπορούν από την πρώτη, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 να κάνουν την αδειοδότηση και ένα άλλο κράτος μέλος είπε ότι για λόγους στρατιωτικής χρήσης δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει την αδειοδότηση για την ζώνη των 800 MHz και αυτό τους το επιτρέπει το άρθρο 1 του προγράμματος για το ραδιοφάσμα. Την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Ραδιοφάσματος συζήτησε με τα κράτη-μέλη και εξηγήσαμε τη διαδικασία παρεκκλήσεως και κάναμε μια έκκληση σε αυτές τις χώρες να μας αναφέρουν εγκαίρως και ταχαίως αν δεν θα μπορέσουν μέχρι το τέλος του έτους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Περνώντα λοιπόν στο άλλο σημαντικό θέμα τη διαδικασία αδειοδότηση, είναι εξίσου σημαντικό να σημειώσουμε ότι προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζοντα τα θέματα αυτά να το κάνουν αυτό διαφανώ και όπου είναι δυνατόν να κάνουν με δημοπρασίες πολυ... με πολλαπλά φάσματα. Όσο πιο πολλά φάσματα είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα, παρέχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και διαφάνεια στου εμπορευομένου. Σημαίνει όμω επίση ότι δεν θα υπάρχει τεχνητό πληθωρισμό των τιμών για τι αδειοδοτήσει που είναι σημαντικό βέβαια, διότι οι πορευόμενοι θα πρέπει να επενδύσουν μεγάλα ποσά για τα δίκτυα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να παράσχουν αυτές τις ε, υπηρεσίες. Λοιπόν, πολυφασματικές δημοκρασίες έχουν προγραμματιστεί 7 φέτος. Είναι κάτι που ενθαρρύνουμε ενεργά. Και αν ένα κάτω μέλος γνωρίζει ότι θα υπάρξει καθυστέρηση για την απελευθέρωση κάποιου φάσματος, κάποιες συχνότητες, δηλαδή 2,6 ε, ή, ε, και 800 MHz θα είναι καλό να δώσουν τι άδειε πρώτα, ώστε οι εμπορευόμενοι να ξεκινήσουν τη δύσκολη διαδικασία ετοιμασία των δικτύων τους. Ε, αυτή η απόφαση ελήφθη σε μια χώρα που ήδη έχει ολοκληρώσει την αντιδότηση του φάσματος 800 MHz παρόλο που το φάσμα, το δίκτυο δεν θα είναι έτοιμο πριν από την Ιανουάριο του 2014. Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο χορηγούνται οι άδειε είναι σημαντικό, Δηλαδή, οι υπάρχουσες άδειε στα 900, 1800 είναι άδειε, στα 800 ή στα 2,6 να διατίθεται στην αγορά και θα πρέπει να υπάρχουν όροι και υποχρεώσεις που επιβάλλουν στους εμπορευόμενου στα κράτη-μέλη. Τα 900 και 1800 αυτό το φάσμα αναφέραμε μια, ότι είναι ο τομέα αναδιάθεση του φάσματος και εκεί υπέχουν υποχρέωση στα κράτη-μέλη ούτω ώστε να επιτρέπουν σε εμπορευόμενου που ήδη έχουν άδειε να δώσουν νέε καινοτόμε υπηρεσίε 4G, θα πρέπει όταν το κάνουν αυτό να μην δημιουργούν προβλήματα για τον ανταγωνισμό για μικρότερε εταιρείε ή για νεοσερχόμενε εταιρείε. Επίση, αν νέε επιχειρήσει, νεοσερχόμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν, θέλουν να εκμεταλλευτούν το νέο φάσμα που διατίθεται, θα πρέπει να επικρατούν οι συνθήκε ώστε οι μικρέ εταιρείε να μπορούν να ανταγωνιστούν, να μπουν στην αγορά και γι' αυτό ενθαρρύνουμε και σε διμερείς επαφέ με τα κράτη-μέλη τα παροτρύνουμε να λάβουν συνδυασμό μέτρων που θα ταιριάζουν κατά περίπτωση ε, στην ιστορία της κάθε χώρας και στην παράση κάθε χώρας αλλά να προσαρμοστούν στις τεχνικές που προτείναμε. Δηλαδή, οι εθνικές αρχές μπορούν να παράσχουν εθνικές υποχρεώσεις ε, περιαγωγής. Ένας μικρός εμπορευόμενος που έφτιαξε το δίκτυό του μόλις τώρα για σταθερό χρονικό διάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από άλλον παλιό εμπορευόμενο με υπάρχον δίκτυο, όριμο δίκτυο, να παράσχει υπηρεσίε μέσω του δικτύου του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άλλο τρόπο για να εξασφαλίσετε την αγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμό είναι επιβάλλοντα ένα όριο στα φάσματα, κυρίω κάτω από το 1 GHz. Από τα 900, στο φάσμα 800 MHz, 900 MHz και έτσι αυτό το περιορισμένο φάσμα που είναι διαθέσιμο να μοιράζεται με τον πιο ακριβοδίκιο τρόπο όσο πιο δίκαια γίνεται, τόσο το δυνατόν περισσότερε εταιρείε να μπορούν να παράσχουν τι καλύτερε ευρυζωνικέ υπηρεσίε που λειτουργούν σε αυτέ τι συχνότητε κάτω από το 1 GHz. Το φάσμα που είναι κάτω από το 1 GHz. Αυτά είναι θέματα που μαζί με τους συναδέλφους στην ομάδα εφαρμογής ε, τα συζητήσαμε. Ήρθαμε σε επαφή με κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η απελευθέρωση του φάσματος και η αδειοδότηση, όλα αυτά γίνονται όσο πιο αμαλά γίνεται, ότι διατίθεται υπηρεσίες στους πολίτες με έναν τρόπο ε, που επιτρέπει τον ανταγωνισμό που θα μειώσει τελικά τις τιμές ε, προς όφελος του καταναλωτού και η οικονομική ανάπτυξη. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ε, κυρία Τσικάου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη διοργάνωση αυτής της ανταλλαγής απόψεων και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση. Είναι πραγματικά κρίμα που δεν είναι περισσότεροι ευρωβουλευτές παρόντες. Θα πρότεινα λοιπόν μετά τις θερινές διακοπές να διοργανώσουμε μία μίνι ακρόαση. Δεν χρειάζεται να είναι τρίωρη, μία μισή ώρα μόνο, μία μίνι ακρόαση όπου θα προσκαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και εκπροσώπους ε, από τα κράτη-μέλη για να μας ε, εξηγήσουν ποιε ήταν οι καλύτερε εμπειρίε του, ώστε να αξιοποιήσουμε τι βέλτιστες πρακτικέ και να δούμε τι προβλήματα αντιμετώπισαν τα κράτη-μέλη και σε τι εμπόδια προσέκρουσαν που τους ε, εμπόδισαν να εφαρμόσουν την οδηγία και γι' αυτό χρειάστηκε παράταση πέραν του της 1ης Ιανουαρίου του 2013 για την απελευθέρωση του ραδιοφάσματος. Θα μπορούσε παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ό,τι αφορά την υποχρέωση περιαγωγής ε, σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ε, τι γίνεται με την υποχρέωση κάλυψης. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικές ε, πρακτικές των κρατών μελών, γιατί κάποιες χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα, θέσπισαν την ε, υποχρέωση κάλυψης για την Ήπεθρο, για τις αγροτικές ζώνες. Από τη στιγμή που εξασφαλίστηκε η κάλυψη στην Ήπεθρο, μπόρεσαν οι πάροχοι να χρησιμοποιήσουν το ραδιοφάσμα και για αστικές περιοχές. Αν μιμούμαστε τη Γερμανία θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ε, και στις δικές μας χώρες πρόσβαση σε όλους τους πολίτες ε, σε ποιοτικέ τηλεπικοινωνίες. Δεύτερη ερώτηση για, το, για την υποχρέωση εθνικού roaming, εθνικής περιαγωγής. Μας είπατε ότι οι νέοι εισερχόμενοι πάροχοι στην αγορά μπορούν να ζητήσουν από έναν παραδοσιακό πάροχο που ήδη είναι εγκατεστημένο στην αγορά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το δίκτυό του για περιορισμένο χρόνο. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Τι εννοείτε για περιορισμένο χρόνο, για πόσο χρόνο δηλαδή. Ευχαριστώ. Α, και έχω και μια τρίτη ερώτηση. Τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, πώς θα μπορούσαμε εμείς να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να τηρήσουν αυτή την προθεσμία και να απελευθερώσουν έγκαιρα το ραδιοφάσμα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ τη συνάδελφη Τικάου. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τικάου. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με τα ερωτήματά σας που αφορούσαν την περιαγωγή. Πράγματι, αυτό θεωρείται ότι είναι ένας μηχανισμός ούτω ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ερχόμενοι ή αυτοί που μπήκαν καθυστερημένα στην αγορά έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν στην παροχή υπηρεσιών ενώ βεβαίως πρέπει να πληρούν υποχρεώσεις να ετοιμάσουν το δίκτυό τους. Και αυτό επιτυγχάνεται πολύ συχνά σε αυτό που αναφέρατε, αυτές τις υποχρεώσεις κάλυψης. Η φύση του ρυθμιστικού μας πλαισίου είναι τέτοια που δεν περιγράφουμε λεπτομερώς στα κράτη-μέλη το πώς θα έπρεπε ή θα μπορούσαν ή πρέπει να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Τους δίνουμε ένα πλαίσιο. Και τα κράτη-μέλη κρίνουν τι είναι ανάλογο και τι είναι ενδεδειγμένο δοθέντων των εθνικών περιστάσεων. Και κυρίως κληρονομιά, όπως αποκαλούμε. Ε, δηλαδή, η κατάσταση ενός μεγάλου κράτους μέλους που ήδη να έχει μεγάλες εταιρείε και ένα μικρό κράτος μέλος που να έχει τρεις εταιρείε, το μεγάλο έχει τέσσερις εταιρείε. άρα διαφέρουν οι καταστάσεις. ακόμα και εντό των παραδειγμάτων υπάρχουν άλλες διαφοροποίησεις. Γι' αυτό θέλαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι με τα κράτη-μέλη. Έχουμε όμως παραδείγματα κατά τα οποία, κατά το παρελθόν, πριν διατεθεί αυτό το νέο φάσμα, ήδη είχαμε ας πούμε την τρίτη, τέταρτη επιχείρηση που ήταν ε, καινούργια εταιρεία που έμπαινε, δεν υπήρχε φάσμα των 900 MHz, μπορούσε να είχε άδεια για τα 1800 MHz ή το φάσμα 3G, το UMTS, στα 2 GHz. Και για να μπορέσουν αυτοί, όταν οι υπηρεσίες 4G ξεκινήσουν, για να μπορέσουν αυτοί, αυτές οι καινούς εταιρείε να αναπτύξουν τη δική τους προσφορά, τις δικές τους υπηρεσίες για τους πελάτες ή αν υπάρχει νέος εμπορευόμενος με άδεια και μπαίνει στην αγορά να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες, θέλαμε η Εθνική Αρχή ε, Αδειοδότησης ή να ζητήσει προσφορά ή να, ζη... επιβάλλει υποχρέωση σε, άλλο σε άλλη επιχείρηση που ήδη έχει άδεια και δίκτυο που καλύπτει όλο το κάτω μέλος να δώσει πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο σε περιοχές όπου η μικρή εταιρεία δεν έχει κάλυψη. Αυτό από μόνο του μπορεί να γίνει παράγοντας που βλάπτει τον ανταγωνισμό. Ε, αν αυτό δεν τέριαζε απόλυτα για να καλύψει τις ανάγκες της μικρής εταιρείας για, μικρή, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γι' αυτό, όπως είπατε, αυτό συνδέεται με τις υποχρεώσεις κάλυψης. Η Γερμανία είναι πολύ καλό παράδειγμα. Γιατί για να εξασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται αυτό το φάσμα για να καλεί τις πιο σημαντικές ομάδες της κοινωνίας και τις πιο σημαντικές περιοχές των κρατών μελών, κυρίως την Ήπεθρο, όπου υπήρχε χαμηλή κάλυψη άλλων ευρυζωνικών υπηρεσιών, κάναν αντίστροφη κάλυψη από ό,τι γινόταν για το GSM. Αντί να ξεκινήσουν από τις πυκνοκατοικημένες πόλεις και να προχωρήσουν από εκεί, επέβαλαν υποχρέωση πρώτα απ' όλα για την κάλυψη των πιο αεροκατοικημένων περιοχών. Και εντός αυτού επιτρέπουν. Όταν να χρησιμοποιηθούν άλλα να χρησιμοποιήσουν άλλα δίκτυα υπό την προπόθεση ότι μπορούσαν να αποδείξουν ότι επένδυαν στην κατασκευή των δικτύων τους στην Ήπεθρο. Αυτό δείχνει το βαθμό της ε, ευελιξίας που διατίθεται στα κάτι μέλη όπου υπάρχουν πραγματικοί κανόνες για το πλαίσιο. Δεν είναι αόριστη εν λευκό επιταγή που δίνουμε στον εμπορευόμενο, πρέπει πραγματικά να αποδείξουν πεδίο στην αγορά και μετά από μια χρονική περίοδο συγκεκριμένη θα πρέπει να μπορούν να παράσχουν οι ίδιες οι εταιρείε αυτές τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ποιο πρέπει αυτό το διάστημα το χρονικό, η αρμόδια Εθνική Αρχή Αδειοδότηση, ανάλογα με τι περιστάσει που κρατούν σε κάθε χώρα, κρίνει. Όσον αφορά το φάσμα και τα όρια στα φάσματα, ε, εκεί τίναμε να εντοπίσουμε σαν βέλτιστη πρακτική ποια είναι, αλλά ακόμα και εδώ αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ε, σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, που υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Αν έχεις τρεις μεγάλες εταιρείες Φερρυπίν, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι καμία από αυτές δεν έχει περισσότερο από, από 20 MHz φάσματος κάτω από το 1 GHz. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό στην άδεια που είχαν για τα 900 και την άλλη που συζητήσουν και πάρουν για τα 800 μεταξύ 800 και 900 σε αυτό το φάσμα συστήσαμε σε κάποιες περιπτώσεις τα κάτι μελη να υπάρχει ένα όριο 20 MHz όσον αφορά τις συχνότητες. Γιατί με τα 20 MHz, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δώσαν αντικειμενικά τεχνικοί, θα μπορέσουν να παράσχουν πλήρες υπηρεσίες μεγάλης ταχύτητας ε, νέας τεχνολογίας. Ενώ άμα χρησιμοποιήσουν ψηλότερο στα 1800 ή στα 2 GHz, εκεί μπορούν να παράσχουν άλλες υπηρεσίες και μπορούν να εξασφαλίσουν και τη συνέχεια των φωνητικών υπηρεσιών που είναι πολύ σημαντικές για όλους τους πολίτες. Πουθενά δεν θα δείτε γραμμένο ότι πρέπει να είναι 20 MHz, ότι θα είναι, πρέπει να είναι λιγότερο ή παραπάνω, διότι πρέπει να ταιριάζει με τις εθνικές ανάγκες. Και κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να μην επιβάλλουν ένα όριο όταν πιστεύουν ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά τους είναι τέτοιος που δεν απαιτείται κάτι τέτοιο ή ότι η κατάσταση είναι αρκετά υγιής, άρα μπορούν ε, επιβάλλοντας άλλες υποχρεώσεις, όπως υποχρεώσεις κάλυψης, ότι μπορούν έτσι να καλύψουν ότι θα διατεθούν ε, παρόμοιες υπηρεσίες σε ανταγωνιζόμενα δίκτυα και καλύπτεται η μεγάλη πλειοψηφία του επικράτειας και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και νομίζω ότι εν αυτή τη ενία κάλυψα τι ερωτήσει σα, Νομίζω ήταν πλήρης, αρκετά πλήρη απάντηση που σα έδωσα. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρο. σα ευχαριστώ για την παρέμβαση και την παρουσίασή σα. Ολοκληρώσαμε το σημείο 22 τη ημερήσια διάταξη. Μπορούμε τώρα να πάμε στο σημείο 23 που αφορά την παγκόσμια διάσκεψη όσον αφορά τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες του Δεκεμβρίου του 2012 στο πλαίσιο της ψηφιακή ατζέντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ε, πολύ έγκυρη αυτή και επίκαιρη πρόσκληση για να σας κάνω μια ενημέρωση για την παγκόσμια αυτή διάσκεψη του Δεκεμβρίου του 2012. Θα διαπιστώσετε και από ε, το έγγραφο που σας μοίρασα ότι βρισκόμαστε σε ένα προκαταρκτικό στάδιο. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια προς το παρόν. Ελπίζω στην πορεία να κατασταλάξουν κάπως τα πράγματα. Απλώς θα σας δώσω μερικά στοιχεία για το τι συμβαίνει, τι είδους θέματα μας απασχολούν, βρίσκονται επιτάπητος και ποια είναι η θέση των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συζήτηση. Καταρχήν, ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, οι παγκόσμιες ε, τηλεπικοινωνίες ε, διαθετούνται σε διεθνές επίπεδο εδώ και καιρό Ήδη από το 1988 έχουμε κανονισμούς για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες και το έγγραφο αυτό βρίσκεται υπό αναθεώρηση τώρα από τα συμβαλόμενα μέρη της παγκόσμιας διάσκεψης. Θα προσπεράσω αυτή την διαφάνεια που μας δίνει το στόχο των, του κανονισμών αυτών που είναι η θέσπιση γενικών αρχών αλλά και θέσπιση κανόνων που εφαρμόζονται από τις διοικήσεις. Θα επανέλθω και στην πορεία της παρουσίασής μου στο θέμα αυτό. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος, ο γενεσιογρός λόγος αυτής της διάσκεψης. Ε, καταρχήν ε, έχουμε την ίδια φύση των ε, τηλεπικοινωνιών, των διεθνών τηλεπικοινωνιών. Η κατάσταση της τηλεπικοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε το 1988. Δηλαδή, τότε είχαμε ε, εθνικά μονοπόλια το 1988, ενώ τώρα έχουμε τον ε, ιδιωτικό τομέα να πρωτοστατεί στις, τηλε, στις ε, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Επίσης έχουμε μετάβαση από τα σταθερά στα κινητά, έχουμε μετάβαση από τη φωνή στα δεδομένα. Οι αλλαγές είναι ρηξικέλευτες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει η αίσθηση ότι ήρθε η ώρα για ανάγκη των κανόνων του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών. Πώς φτάσαμε τώρα στην παγκόσμια διάσκεψη. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε τελευταία στιγμή λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Πολλά ψηφίσματα έχουν υιοθετηθεί το 2010 αποφασίστηκε ότι ήρθε πια η ώρα να οργανωθεί αυτή η παγκόσμια διάσκεψη για μια σοβαρή πια αναθεώρηση των κανονισμών για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Μάλιστα αυτή η διαδικασία, αυτό το εγχείρημα εμπίπτει σε ένα πλαίσιο εγχειρημάτων. Βλέπετε εδώ ε, διάφορα ε, επιχειρήματα που τα βλέπουμε και στο ίντερνετ και στις, ε, στους κανονισμούς. Πολλές συζητήσεις γίνονται παράλληλα και προσπαθούμε ε, να τις παρακολουθήσουμε ώστε να έχουμε μια συνεπή προσέγγιση, κάτι που δεν είναι εύκολο πάντα. Πάντως είναι σημαντικό η φιλοσοφία ε, που υιοθετούμε είναι καταστελεγμένη και τεκμηριωμένη, γιατί δεν έχουμε μία και μόνο οντότητα. Έχουμε το Φόρουμ για τις Παγκόσμιες Τηλεπικοινωνίες, υπάρχει το ITU και σας έδωσα εδώ τα ακρονίμια. Μπορεί να μην ξέρετε ότι τα μισά περισσότεροι από εσάς αλλά πολλά συμβαίνουν. Το πληρεξούσιο, υπάρχουν, υπάρχει το ICAN, CCT, πολλές συζητήσεις γίνονται παράλληλα σε διάφορα φόρα για τα θέματα αυτά. Ποιοι είναι τώρα οι συμμετέχοντες οι φορείς. Βλέπετε είναι αρκετά μικρά τα γράμματα, αλλά μην ανησυχείτε, θα σας μοιράσω και ε, κείμενο. Έχουμε τα κράτη-μέλη. Φυσικά στο, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν έχουμε μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κράτη-μέλη αποκαλούνται από την διάσκεψη και τα μέλη της διάσκεψης της ITU. Είναι τα συμβαλόμενα μέρη κατά κάποιο τρόπο, όχι τα κράτη-μέλη. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ των μελών ε, της ITU και των ε, υπογραφών ε, των κανονισμών. Υπάρχει μια επικάλυψη, αλλά δεν ταυτίζονται οι δύο έννοιες. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση, να υποβάλουν προτάσεις ε, με διαφορετική ιδιότητα βέβαια και καθεστώς από ό,τι τα κράτη-μέλη, αλλά και η κοινωνία των πολιτών μπορεί να μεταφέρει τη γνώμη της και είναι πολύ σημαντικό να το τονίζουμε ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη και ε, υπογράφουν ε, τους κανονισμούς για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες και μάλιστα αργότερα θα προσχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα. Ένα από τα ενδιαφέροντα φαινόμενα που βλέπουμε και θα σας ε, ενημερώσουν για τις, ε, τις προετοιμασίες ε, για το ραδιόφάσμα, πολλές, σημασίες, πολλές προετοιμασίες γίνονται σε μια ομάδα γιατί έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, 150 και εκεί είναι πολύ δύσκολο να τις διαχειριστούμε. Και υπάρχει και η ITU που έχει τη γραμματεία της, διαδραματεί σημαντικό ρόλο, αλλά φυσικά το βασικό είναι τα μέλη της. Έχουμε τρία είδη ερωτήσεις, ε, προτάσεων που φτάνουν σε αυτή την παγκόσμια διάσκεψη. Υπάρχει ε, ε, ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την ITU που καταρτίζει ένα έγγραφο που βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης και που περιλαμβάνει ένα συμπίλημα, ένα συγκερασμό όλων των προτάσεων που γίνονται. Έχουμε περιφερειακές ομάδες. Έχουμε την, Ευρωπαϊκή Ομάδα Ενδιαφέροντος και αυτοί που βάλουν προτάσεις. Όλες αυτές οι προτάσεις θα συμπληθούν. Υπάρχει τεράστιο χαρτομάνι, πάντως ε, ως προς το περιεχόμενο, μία-δύο εβδομάδες πριν την παγκόσμια διάσκεψη θα έχουμε και νέε προτάσει. Γιατί δύο εβδομάδε πριν την διάσκεψη λίγη η προθεσμία για τι ε, τροπολογίες και τι προτάσει. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι για μερικέ τουλάχιστον εκπλήξει όσο πλησιάζει η μέρα της παγκόσμιας διάσκεψης. Τώρα, ποια είναι, ποιες είναι οι προτάσεις στο περιεχόμενό τους, τους ε, τις συνοψίζω με κάπως νομικούς όρους. Αυτό είναι το είδος ε, των θεμάτων που καλύπτουν οι προτάσεις. Αφορούν περιαγωγή, κατάχρηση, απάτη, φορολογία, τη την αδιαφάνεια των διαδρομών, γενικά οικονομικά ζητήματα, όπως ποιος πληρώνει γιατί και πώς μπορούμε να αποκομίσουμε κάποια χρήματα από τις τηλεπικοινωνίες, διαφοροποιημένη διαχείριση ροής, οργάνωση όλων αυτών, γιατί η κίνηση, η ροή στο ίντερνετ είναι προ όλε τι κατευθύνσει. το θέμα τη κυβερνοασφάλεια και η καταπολέμηση των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Είναι μη εξαντλητικός αυτό ο κατάλογο, αλλά τέτοιου είδου ζητήματα καλύπτονται στι προτάσει. Τώρα, Ποιε είναι οι συζητήσει που είχαμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με του εταίρου μα, όπω τη Ρωσία ή την Τουρκία. Καταρχήν είπαμε ότι πρόκειται για μια ε, συνθήκη από 10 άρθρα, 40 ε, σελίδες ε, και πρόκειται για μια αναθεώρηση μιας, σελί... μιας συνθήκης με 60 σελίδες, με πολύ περισσότερα άρθρα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της συνθήκης, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε την αναθεώρηση σε επίπεδο βασικών αρχών. Και φυσικά η έκβαση θα πρέπει να είναι ουδέτερη και από τεχνολογική άποψη και άποψη αγοράς. Γιατί θα ήταν δυσάρεστο να αρχίσουμε ρυθμίσεις για με βάση την σημερινή τεχνολογία ή την πρόσφατη τεχνολογία και να αποκλείσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις που κατά πάσα πιθανότητα θα λάβω χώρα πολύ σύντομα. Οπότε είναι σημαντικό η συνθήκη να, να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Το θέμα της ασφάλειας είναι ένα βασικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη δεν είναι κατά ε, ενός πιο ασφαλού συστήματος τηλεπικοινωνιών. Αλλά ούτως ή άλλως θα το κάνουμε. Θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να μας λένε ότι θα πρέπει να είναι ασφαλής η τηλεπικοινωνίες. Όχι, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς στα πλαίσια των δικών μας κυρίαρχων δικαιωμάτων. Και συνήθως ε, στον τύπο ε, αναφέρονται διάφορα για το διαδίκτυο και η συζήτηση δεν είναι σαφής, γιατί το θέμα δεν είναι αν λέμε ναι ή όχι στο διαδίκτυο, γιατί ούτως ή άλλως το διαδίκτυο χρησιμοποιεί τις γραμμές των τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει μια άλλη επίδραση. Πάντως είπαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επέκταση της ηθίκης ε, για κάθε ζήτημα που αφορά το διαδίκτυο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης ένα χαρακτηριστικό επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που συμμερίζουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε μετά το Ντουμπάι να γυρίσουμε και να πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε το πακέτο μας ή το κοινωτικό μας κεκτημένο. Το κοινωτικό κεκτημένο θα πρέπει να παραμείνει άθικτο. Τώρα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι του όλου εγχειρήματο. Ο πρώτος κίνδυνος είναι Όπω είπα και προηγουμένω για τι κατευθυντήριε γραμμέ, ο κίνδυνο είναι να μην κάναμε σωστά το έργο μας ε, ε, και να υπάρχει συμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό το απευχόμαστε και θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε να αποφύγουμε μια τέτοια συμβατότητα. Επίσης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά κανόνων και διατάξεων που περιορίζουν τη χρήση του διαδικτύου και τον καινοτόμο χαρακτήρα των τεχνολογιών ουσιαστικά δηλαδή στο μόνο ή περιορίζουν την καινοτομία, αυτό δεν το δεχόμαστε. Η ουδετερότητα του δικτύου είναι αυτονόητη η ανάγκη ουδετερότητας του δικτύου. Έχουμε τέτοια πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θεμελιώδες για μας ζήτημα. Υπάρχει κίνδυνος όμως να επηρεαστεί και η ουδετερότητα. Και κάτι που ανέφερα ρητά εδώ, στις διαπραγματεύσεις αυτές πολύ συχνά ε, διαβάζουμε κάπως ασαφή κείμενα. Δεν είναι κείμενα ευανάγνωστα που δεν επιδέχονται παρερμηνίας. Δυστυχώς είναι κάπως ασαφή τα κείμενα, οπότε καθένας μπορεί να τερμινεύει με διαφορετικό τρόπο. Αυτός είναι σημαντικός κίνδυνος. Να έχουμε δηλαδή στις διαπραγματεύσεις κείμενα που θα είναι ευανάγνωστα και σαφή και να μην επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες. Γιατί χωρίς τέτοια σαφή κείμενα υπάρχει κίνδυνος να κατακαιρματίσουμε το διαδίκτυο με διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, κάτι που θα αποβεί βάρος φυσικά των τηλεπικοινωνιών. Όπως είπα και προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, πολλές διαφορές ε, μεταξύ του 2012 και του 1988. Και φυσικά έχουμε αντίστοιχα νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πολύ πιθανό πολλά από αυτά να επηρεαστούν από τις συζητήσεις ε, της παγκόσμιας διάσκεψης για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Φυσικά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει γιατί δεν θα είναι ανώδυνη για τις ε, νομοθεσίες της αυτή η διάσκεψη. Και φυσικά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι τμήμα του ε, και ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ομάδας αλλά και της παγκόσμιας οπότε θέλουμε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο στην παγκόσμια συζήτηση και να φανούμε ως ενισχυμένη, ε, δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο ρόλος Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει τονιστεί η σημασία της ενιαίας φωνής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ενιαίας δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι συμβαλόμενο μέρος, δεν έχει υπογράψει ξεχωριστά τη συνθήκη. Συμμετέχουμε σε όλες τις συνεδριάσεις που μας αφορούν και μπορούμε να λάβουμε και το λόγο, αλλά σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη του ITU. Και αυτό μερικές φορές περιπλέκει τα πράγματα, το προσπαθούμε να προβάλλουμε την κοινοτική άποψη. Το άρθρο 218 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τη διαμόρφωση κοινή θέση για θέματα που εμπίπτουν στην κοινοτική νομοθεσία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση σχετική στο Συμβούλιο. Δεν έχει ακόμη εγκριθεί, δεν έχει οριστικοποιηθεί η πρόταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπή, οπότε δεν μπορώ να επεκταθώ στο περιεχόμενό τη. Πάντως ε, γίνεται αυτή η προετοιμασία ώστε να υποβληθεί μια ενιαία θέση, ενιαία προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια διάσκεψη του Δεκεμβρίου. Οπότε θα πρέπει να έχουμε έγκυρη προετοιμασία, συζητήσεις με πολλούς ενδιαφερομένους, με κράτη-μέλη, με τη βιομηχανία, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ώστε να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση και κοινή αντίληψη για το πού μας οδηγεί αυτή η διαδικασία και ποια έκβαση επιθυμούμε. Γι' αυτό και προετοιμαζόμαστε εγκαίρως ώστε να ε, λειτουργούμε ομαλά και συνεργαζόμαστε και με την ομάδα του Ντουμπάι και την ομάδα των Βρυξελών ώστε να αποτρέψουμε τους κινδύνους που σας παρουσίασα προηγουμένως. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Προσπάθησε την πρώτη παρουσία μου να την ε, κρατήσω σε ένα σχετικά γενικό επίπεδο. Πάντως θα απαντήσω και πιο λεπτομεριακά στο μέτρο που θα υποβληθούν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Η κυρία Ούμπνερ έχει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ. Η παγκόσμια διάσκεψη του Δεκεμβρίου φαντάζομαι δεν θα καλύψει όλα αυτά τα θέματα που μας ε, περιγράψετε γιατί ε, όλα αυτά τα θέματα που μας είπατε καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα και ίσως το σύνολο των δραστηριοτήτων ε, ε, της Επιτροπής ή αυτής της ομάδας, της Ένωσης που δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή αλλά έχει και ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο θέμα, στο μήνυμα της διάσκεψης του Ιανουαρίου. Δηλαδή έγινε κάποια ανταλλαγή απόψεων για την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες αν το δίκαιο είναι σαφές ή όχι. Ποια είναι τα συμπεράσματα της ε, διάσκεψης και ποιο ήταν το κυρίως θέμα. Μιλήσατε για όλα τα θέματα, επικεντρωθήκατε στα πάντα ή επικεντρωθήκατε σε δύο-τρία κυρίως θέματα και ε, ανταλλάξατε απόψεις για την τεχνολογία, για την πρόσβαση στην τεχνολογία, γιατί συμμετείχαν και εξωκοινωτικές χώρες στη διάσκεψη αυτή και οι διάφορες διατάξεις είναι αντιληπτές και βανάγνωστες για όλους. Σα ευχαριστώ. Μας ευχαριστώ κύριε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν επίσης για την παρουσίασή του. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. γιατί μπορεί να είναι αόρατες οι τηλεπικοινωνίες, αόρατο και άχρο το διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά είναι το καλύτερο εργαλείο για τη μελλοντική ανάπτυξη σε οικονομικό επίπεδο. Το Σεπτέμβριο, ίσως και αργότερα, θα λάβει χώρα πάλι μια τέτοια παρουσίαση και ελπίζω ότι θα μπορούσατε σε αυτή την περίπτωση να μας δώσετε και πάλι τα φώτα σας, να μας δώσετε κάποια στοιχεία από την παρουσίασή σας εν ώψη αυτής της συνάντησης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς και να καταλάβει ακόμα περισσότερο όλες τις πτυχές αυτού του δύσκολου θέματος. Είμαι σίγουρη όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερα σε σχέση με τα θέματα αυτά, γιατί σε τελική ανάλυση εμείς θα πρέπει και εμείς να παίξουμε κάποιο ρόλο για τη διαμόρφωση αυτού του τομέα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο α, ακόμα χωρίς ε, ρύθμιση θέματα στην Ευρώπη και πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να συγκεντρώσουμε αρκετέ γνώσεις για να μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να βρούμε τη βέλτιστη λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη της. Γιατί αλλιώς αυτά τα οποία βλέπουμε σε επίπεδο οφθαλμοφανές δεν είναι αυτά τα οποία προσδιορίζουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Είναι τα αόρατα στοιχεία που το κάνουν. Η Αμέλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία αυτή να λάβω το λόγο. Προφανώς το Δεκέμβριο στη συνδιάσκεψη θα υπάρχει ευρύ πεδίο του επιστητού που θα αντιμετωπιστεί, αλλά υπάρχει και ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο μένει έξω από αυτές τις διαπραγματεύσεις της διεθνούς Ένωσης τη τηλεπικοινωνία, είναι η κοινωνία των πολιτών η οποία εμποδίζεται από το υψηλό κόστος <clears throat> συμμετοχής να λάβει μέρος στα τεκτενόμενα και επίσης επειδή δεν έχει πρόσβαση στην τεκμηρίωση και ουσιαστικά σε όλη τη διαδικασία που οδηγεί στα συμπεράσματα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών προβλέπει η Κομισιόν το Δεκέμβριο να κάνει κάτι για να ευνοήσει τη συμμετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών το Δεκέμβριο και στη διάσκεψη αυτή και σε μελλοντικέ εκδηλώσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Πώς προβλέπει η Κομισιόν να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο λοιπόν για να δώσετε απάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις αφορούσαν τη συμμετοχή και τη διαδικασία. Σημαντικές ερωτήσεις, σημαντικά θέματα που δεν τα τόνισα αρκετά. Αυτό επί δύο-τρία χρόνια γίνεται και εμφανίζονται προτάσεις κάποιες σοβαρότερες από άλλες, άλλες αφέστερες από τις άλλες. Επί του παρόντος διεξάγεται συζήτηση με θέμα τη διαφάνεια της διαδικασίας του ε, ITU και είναι πολύ σημαντικό ε, και πολύ στεναρά Ευρώπη ζήτησε από τη Γραμματεία του ITU να διεξαχθεί σωστά ε, η διαδικασία και να διαθεθεί δημοσία το έγγραφο το οποίο θα είναι το προϊόν. Να, το δουν και άλλες χώρες του κόσμου. Δεν τόσο διαφανεί όπως τα κρατημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό και θα πολεμήσουμε, θα δώσουμε τη μάχη ούτως ώστε τα βασικά έγγραφα να διατίθενται σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά τη συμμετοχή των εταίρων, ανέφερα την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει σε επαφή με τους εταίρους, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι εντελώ διαφανής η προσέγγιση. Αν βλέπω τους παρόντες στη Γενέβη και τις οργανώσεις που εκπροσωπούνται εκεί, καλύπτεται ένα αρκετά ευρύ φάσμα, αντίθετα από ό,τι είδαμε σε κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και όλες οι αντιπροσωπείες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. Είμαστε υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας βέβαια. Στην πράξη πιθανότατα όλοι μπορούν να έχουν τα έγγραφά τους μέσω των διαφόρων οργανισμών που συμμετέχουν. Πρωτιθέμεθα στην προπαρασκευή μας προς το Wikit του Δεκεμβρίου να έρθουμε σε επαφή με το Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερομένους και ίσως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορούμε να επανέλθουμε. Το προσφέρατε, με τα χαράς δεχτούμε την προσφορά σας με ευρύτερη συμμετοχή, ευρύτερο πλαίσιο, ακροάσεις, ότι θέλετε να διοργανώσετε. Είναι σημαντικό και με τα χαράς να συμμετάσχουμε στη μάχη και να μοιραστούμε τη γνώση που διαθέτουμε μαζί σας και με τους Ευρωπαίους εμπορευαμένους και ενδιαφερομένους ε, και έτσι θα πάρουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες προετοιμαζόμενοι για την εκδήλωση. Και συμφωνώ ότι πράγματι πρέπει να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών. Ήδη μιλήσαμε με κάποιους φορείς κοινωνίας των πολιτών, γνωρίζουν το θέμα. Καλό δημόσιο ε, έγγραφο παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, όπου δίνει μια γεύση αυτό το έγγραφο τα είδη των θεμάτων που συζητούνται. Το άλλο το ερώτημα για τα διάφορα ζητήματα δεν έχει αποφασιστεί τίποτα, το ξεκαθαρίσουμε. Μία γεύση σας έδωσα όσον αφορά την φύση των προτάσεων που γίνονται. Άλλες είναι πιο σοβαρές, άλλες λιγότερο. Πρέπει όλες να εξεταστούν. Η αδίποτε υποβληθεί σαν πρόταση θα συζητηθεί και θα συζητηθεί και θα χωνευτεί ούτως πίν στη διασκεψή. Σε αυτή τη φάση δεν έχουμε κανένα συμπέρασμα. Κάποιες προτάσεις είναι πολύ γενικέ. Ε, υψηπετείς αρχές που δεν ξέρουμε τι σημαίνουν, άλλες είναι λεπτομερέστατες, εμπεριέχουν τεχνικά σφάλματα, δεν ταιριάζουν με κάποιες νομοθεσίες, άρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν, άρα είναι ένα μείγμα προτάσεων που έχουμε και θέλουμε να δημοσιοποιηθούν όλες οι προτάσεις και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας κάποιες λεπτομέρειες των θεμάτων που συζητούνται. Όπως προανέφερα, η διαδικασία δεν είναι αυτή που συνηθιζόταν με το WRC όπου είχατε την πρόταση που συζητείτε για δύο χρόνια γίνονται τεχνικές μελέτες και μετά υποβάλλετε και συζητείτε περαιτέρω. Μπορεί να έρθουν και προτάσεις δύο τις εβδομάδες πριν από τη διάσκεψη και οι αντιπροσωπείες μετά θα πρέπει να τις συζητήσουν. Ίσως είναι οι πιο περίπλοκες διαπραγματεύσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει μέχρι τώρα λόγω της ελήψεως συνεπούς καλής προετοιμασίας αν θέλετε. Έχουν την προετοιμασία διάσκεψης και στη διάσκεψη θέλουμε να υπάρχει καλή ροή πληροφοριών και να μην φύγουμε από την διάσκεψη βλέποντας να αναφύονται κάποιες εκπλήξεις μετά. Ευχαριστώ. Καλώς, σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβασή σας. Περνάμε στο σημείο 24 της ημερήσιας διάταξης που είναι και η τελευταία παρουσίαση που αφορά την επικείμενη δέσμη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Κάλμπερ θα μιλήσει και το δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα θα σας παρουσιάσω τη θέση μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στατική για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Εκπροσωπώ τον Τζουζέ Πελαμόντε, τον επικεφαλής της μονάδας που ηγείται τη τους. Δυστυχώς δεν μπορούσε να παρίσταται σήμερα το απόγευμα. Εντάχει, ας πούμε, παρουσιάσουμε το θέμα. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Είδαμε στον τύπο μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στο διαδίκτυο, σε ιδιωτικά στοιχεία, σε συστήματα ασφαλείας. Και η οικονομία μας και η κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις προόδους που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Είδαμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αν το διαδίκτυο χρησιμοποιεί το περισσότερο σε όλη την Ευρώπη αν οι χρήστες το εμπιστευόταν περισσότερο και φοβόταν λιγότερο για την ασφάλεια. Πέρα όμως ε, από τη συμπεριφορά μας σαν άτομα ε, και κινδυνεύουν όμως και οικονομίες, εθνική ασφάλεια. Ε, και αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Οικονομία. Και το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο. Δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν έχουμε ένα εθνικό νησί ευρωπαϊκό νησί. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η στατική για τον κυβερνοχώρο χρειάζεται σφαιρική προσπάθεια των διαφόρων υπηρεσιών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη Επιτρόπου Κρούς, από την DG Connect, από την Επίτροπο Μάλστρομ και την Αντιπρόεδρο Άστον της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτές είναι οι τρει υπηρεσίε που καταβάλουν προσπάθειε όσον αφορά τη διαμόρφωση αυτή τη στρατηγικής για τον κυβερνοχώρο. Τώρα, να σας δείξω ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θέλουμε να έχουμε ασφαλές περιβάλλον που δημιουργεί εμπιστοσύνη, που προωθεί τις βασικές αξίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρώπης. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες, κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των δικτύων επικοινωνιών, των υποδομών, των εφαρμογών. Πέρα από αυτό όμως, θέλουμε να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Αυτή είναι η άλλη διάσταση. Έγκλημα στο κυβερνοχώρο. Υπάρχουν εκτιμήσεις Ε, η αξία, οικονομική αξία των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο φτάνει στα επίπεδα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Δεν ζούμε σε νησί, όπως σας είπα. Άρα, χρειάζεται συντονισμένη η δράση. Συγχρονισμό όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, συνεργασία και με τους εταίρους μας ε, εκτός της ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ποιε είναι οι βασικέ δράσει που θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη στρατηγική την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν τις δυνατότητες να προστατεύσουν τα δίκτυά τους, τις υποδομές τους, τους χρήστες, τους πολίτες, ότι μπορούμε να αντιδράσουμε όχι μόνο σε εθνικό, αλλά συνεκτικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν υπάρξουν κάποιες επιθέσεις, κάποιες υποθέσεις που ξεπερνούν ένα κράτος μέλος, να υπάρχει μηχανισμός συνεργασίας για να προστατεύονται οι γειτονικέ χώρε εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αλλά να μην λησμονούμε ότι οι πληροφορίε και η τεχνολογία επικοινωνία και το διαδίκτυο παίζουν πολύ σημαντικό οικονομικό ρόλο, διευκολύνουν το επιχειρήν, δημιουργούν επιχειρήσει, οπότε έχουμε και σαφή διάσταση εσωτερική αγορά. Θέλουμε λοιπόν να αρπάξουμε την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή αγορά να αναπτυχθεί αυτή η αγορά, να είναι ασφαλή η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται και ασφαλή η λύση που βρίσκουμε. Πέρα από την πτυχή της αγοράς και την πτυχή του χρήστη και αυτή τη διάσταση, δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτές, ε, αυτές οι κλιματικές πράξεις και αν μας συμβούν θέλουμε να μειώσουμε τι συνέπειε των πράξεων αυτών. Ε, θα πρέπει οι δυνάμεις της τάξης να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους επιθέσεις. Ερωτήσεις. Πώς ε, μπορείς να βρεις στοιχεία ε, που να μπορούν και αποδεικτικά στοιχεία ενός αδικήματος, ενός εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία σε δίκη. Μπορούμε να κάνουμε πολλά όσον αφορά την ασφάλεια. Τα ξεκινούμε από το χρήστη πρώτα απ' όλα. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι χρήστες. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ε, χρήστες και τις εταιρείες ο καθένας να γνωρίζει πώς να προστατευτεί, πώς να κινείται στο διαδίκτυο, πώς να μειώνει τους κινδύνους, πώς, πώς να είναι ασφαλής ερευνώντας και ανοιχνεύοντας το διαδίκτυο και ωφελούμενος στο διαδίκτυο. Ε, είναι σαν την ε, εξέλιξη στον τομέα των ε, όπλων εδώ και εδώ προχωρούμε. Είναι σαν ένα είδος αγώνα η πρόοδος τεχνολογίας είναι σαν να συναγωνίζεται με κάποιον σε, σε, καινούργια όπλα. Πρέπει να είσαι πιο γρήγορο από αυτό που μπορεί να επιτεθεί. Και γι' αυτό προβλέπουμε μια στρατηγική για να αυξήσουμε τι επενδύσει ε, στην έρευνα, αλλά όχι μόνο αυτό, όχι μόνο σε απόλυτες τιμέ, αύξηση τη επένδυση, αλλά να δούμε πώ μπορούν να είναι καλύτερε οι προσπάθειε στην τεχνολογία και να καλύπτουμε καλύτερα τι ανάγκε που υπάρχουν τη κοινωνία των κρατών κλπ τις τεχνολογικές. Ε, υπάρχει διεθνής διάσταση της ασφαλείας στο κυβερνοχώρο. Εκεί συζητούμε με τους ομολόγους μας θέματα κοινών συμφερόντων που ξεπερνούν τις εθνικές ε, ανησυχίες. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε, να αποφύγουμε επιθέσεις που προέρχονται εκτός συνόρων Πώ μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίε, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία με τους ομολόγους μας σε όλο τον κόσμο και μετά πού βρισκόμαστε όσον αφορά την προετοιμασία της στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει νομοθετικού περιεχομένου πρόταση που θα εδράζεται επί του άρθρου 114 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης βασικά. Τρεις θα είναι οι βασικοί άξονες. Πρώτον, να αυξηθούν οι εθνικές δυνατότητες, να υπάρχει ετοιμότητα, αποτελεσματική ανταπόκριση σε οδήποτε γεγονός ή επίθεση. Θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να διορίσουν εθνική αρχή που θα είναι αρμόδια για την εμπετόπιση αυτών των γεγονότων και όμως που θα έχει το δικαίωμα να συζητεί με αντίστοιχες, ε, σε αντίστοιχους άλλα κράτη-μέλη. Θα δημιουργήσουμε πλαίσιο συνεργασίας ε, όπου θα γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών σε κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ αρμοδίων αρχών και διαφόρων μηχανισμών αμυντικών των χωρών μελών, να υπάρχει καλή προστασία κατά ε, γεγονότων, επεισοδίων που ξεπερνούν την ευρωπαϊκή κλίμακα, κατά επιθέσεων τέτοιων και θέλουμε να συμμετάσχει και ο ιδιωτικό τομέα, να είναι πιο έτοιμο ο ιδιωτικό τομέα, να αυξήσει το επίπεδο προστασίας του και έχουμε και τη διάσταση αγοράς, να προωθήσουμε τη διαχείριση του κινδύνου όπου η προστασία των συμφερόντων, ε, η προστασία των εταιριών γίνεται τμήμα της νοτρο... κομμάτι της νοτροπίας εταιρείας. Και ενημερώνει αν δεχτείς κάποια επίθεση σαν εταιρεία και αν δημιουργηθούν κάποιε ζημίε και δεν έχει κάνει κάτι, μπορεί να θεωρηθεί ότι είσαι υπεύθυνη σαν εταιρεία και μπορεί να ζητηθεί να καταβάλει αποζημιώσει. Αυτά και σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Αντεστότερ. Κύριε Αντεστότερ. Uh, σα ευχαριστώ. Έχω λίγα μονάχα ερωτήματα προς την Κομισιόν σε σχέση με τη μελλοντική στρατηγική στον κυβερνόχωρο τι είδους διαχωρισμό των διαφορετικών πτυχών της στρατηγικής για τον κυβερνόχωρο προβλέπετε. Μία στρατηγική θα αναπτύξετε για όλα τα οποία μπορούν να μπουν μέσα στον χώρο των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος διαχωρισμός μεταξύ των μέτρων διαφύλαξης όταν έχετε να κάνετε με υλική υποδομή όπως είναι τα καλώδια και άλλου είδους ε, στοιχεία όπως είναι η πληροφορία διαμετακομισμού και περιεχόμενο χωριστά. Αν θα έχετε λοιπόν μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση για τις διάφορες, τους διάφορους τομείς προστασίας. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο η εκτίμηση κινδύνου που ζητάτε για τις ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να επεκταθεί και σε εταιρείε δημοσίου συμφέροντος αν θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφόρηση και αξιόπιστα και ανθεκτικά συστήματα για τη μετάδοση των πληροφοριών ή αν απλώς περιορίζεστε σε αξιολόγηση κινδύνου για ιδιωτικές εταιρείες, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ε, υποδομής είναι στα χέρια ιδιωτικών εταιρεών. Αν η Κομισιόν θέλει να προασπίσει και το δημόσιο συμφέρον, αυτό θα είχε πολύ ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ. Κυρία Ήπνερ. Ευχαριστώ. Το σημερινό θέμα, παρά τα φαινόμενα, είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον μας. Το διαδίκτυο είναι καταπληκτική εφεύρεση, αλλά ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνο όπλο, ιδιαίτερα αυτά σε χέρια κακοπροαίρετων που μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές. Επίσης, ε, είναι η πολυεπίπεδη η ανάγκη ασφάλειας στο διαδίκτυο. Πολλοί προσπάθησαν να, ε, να υπεξαιρέσουν χρήματα από τραπεζικού λογαριασμού. Είναι ένα πρώτο επίπεδο. Αλλά υπάρχει θέμα ε, και διεθνούς, εθνικής ή διεθνούς ασφάλειας, γιατί το διαδίκτυο δεν γνωρίζει σύνορα. Οπότε το θέμα της ε, διεθνούς ασφάλειας και η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των χωρών είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Το ίδιο σημαντικό είναι και η ανάληψη δραστηριοτήτων για να αποτραπούν τέτοιοι κίνδυνοι. Το διαδίκτυο μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες ε, από δημόσιες αρχές. Μπορεί να καταστρέψει ζωές δηλαδή. Μπορεί το, τέτοιου είδους πληροφορίες να γίνουν όπλο στα χέρια άλλου ανθρώπου πολλά εγκλήματα μπορούν να γίνουν μέσω του ίντερνετ. Επίσης, ε, μέσω του ίντερνετ διαπράττονται και σεξουαλικά εγκλήματα. Ε, δεν είναι κάτι δηλαδή περιορισμένο. Γιατί, επαναλαμβάνω, μια και τα γνωρίζει σύνορα μπορεί να φτάσει σε μια διεθνή διάσταση ένα τέτοιο έγκλημα. Οπότε η διαπαιδαγώγηση και η αποτροπή αυτών για την αποτροπή αυτών των κινδύνων θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη από το νηπιαγωγείο και το σχολείο. Πρόκειται ε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως σας είπα. Μας είπατε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα εγκλήματα, να τα προλάβουμε επίσης αν γίνεται, να δώσουμε μια έμφαση στην πρόληψη. Πιο... Τι γίνεται όμως ε, σε περίπτωση που εξαφανίζονται, που σβήνουν κάποιες σελίδες που δεν έχουν καν θέση στο ίντερνετ. Ε, ποια υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης ώστε να αποσύρονται αυτές οι σελίδες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχετε δυνατότητα άμεσης δράσης, ώστε αμέσως να κλείνετε τέτοιες σελίδες. Ώστε να μην χρειάζεται να ακολουθεί μια χρονοβόρα διαδικασία προκειμένου να αφαιρεθούν ή να φραχθούν σελίδες στο ίντερνετ που ούτως ή δεν έχουν θέση εκεί. Είναι σημαντικό το θέμα τη άμεση αντίδραση, αλλά ποιο είναι ο χρόνο αυτή τη αντίδραση Υπάρχει τέτοια δυνατότητα πραγματικά άμεση αντίδραση, ώστε αμέσω να μπορεί κανεί ε, σε περίπτωση που διαπιστώνει ύπαρξη τέτοιου σελίδα να τι ε, αποσύρει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την παρέμβαση. Για τα συμπεράσματα, ο κύριος Κάλμπερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Um, uh, Να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Η στρατηγική κυβερνασφάλειας δεν μπαίνει σε τεχνικό επίπεδο σε διάφορες τεχνολογίες, το πώς λειτουργούν διάφορες εφαρμογές, διάφορα στρώματα υποδομής, διάφορες στρώσεις υποδομής πώς πρέπει να προστατευθούν. Θέλουμε απλώς όλες οι εφαρμογές συστήματα και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα έχουν εφαρμοστεί θα, είναι, να πρέπει να είναι ανάλογα με τους κινδύνους που αφορούν αυτό το, το μηχάνημα ή το τμήμα του λογισμικού κτλ. Και όχι να έχουμε πολύ δάπανες λύσεις οι οποίες ξεπερνούν το επίπεδο αυτό, το αναλογικό. Ο στόχος μας λοιπόν είναι μια γενική αύξηση του επίπεδου ασφαλείας και το να εξασφαλίσουμε ότι σε κάθε σε κάθε επίπεδο, σε κάθε στρώση από, το τερματικό, ε, από την τερματική συσκευή που έχετε μέχρι το δίκτυο, μέχρι τη φυσική υποδομή υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια και ο κάθε εμπλεκόμενος θα πρέπει να παρέχει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στο κομμάτι αυτό της αλυσίδας για το οποίο είναι υπεύθυνο. <clears throat> σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου τώρα, το ερώτημά σας είναι ιδιαίτερα έγκυρο. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να είναι χωρίς διακοπή η ασφάλεια και ότι εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος είναι στον ασθενέστερο κρίκο. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του και να παίξουν όλοι το ρόλο τους. Φυσικά οι μεγάλες εταιρείε πρέπει να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο και ο δημόσιος τομέας επίσης, αλλά όταν η παροχή μιας υπηρεσίας, η λειτουργία μιας υπηρεσίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κάποιους χρήστες, κάποιες εταιρείες ή κάποια άτομα ή τη σύνολη κοινωνία, αυτός ο οποίος ελέγχει το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχει τη σωστή διαχείριση κινδύνου και παίρνει τα κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για να υπάρξει μείωση του κινδύνου. Τέλος, για το θέμα της ταχείας αντίδρασης μέσα στα σύνορά μας, για να ε, αφαιρέσουμε εκκληματικού περιεχομένου ιστοσελίδες που έχουν αναρτήθει. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που το αντιμετωπίζει η στρατηγική μας σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειες. Γιατί η δράση για να κλείσει κανείς μια ιστοσελίδα εξαρτάται από τις ε, διοκτικές αρχές και τα δικαστικά συστήματα της κάθε χώρας αυτό το οποίο χαιρετίζουμε από τη δική μας πλευρά είναι να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός συντονισμός, ώστε όταν μια χώρα αναφέρει μια εγκληματική ιστοσελίδα σε μια άλλη χώρα, τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός με τον οποίο η άλλη χώρα μπορεί να κάνει τα κατάλληλα βήματα για να εξαλειφθεί αυτή η ιστοσελίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν εδώ μέχρι τώρα. Ολοκληρώσαμε τα σημεία της στη διάταξη, ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Επιτροπής, ε, ραντεβού στις 3 Σεπτεμβρίου του 2012, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Καλό καλοκαίρι, καλές διακόπες, ευχαριστώ.